με το Spitzenkandidat, αλλά είμαι υπερήφανη που όλα τα βασικά θέματα για τα οποία αγωνιστήκαμε πλέον εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω σοσιαλδημοκράτε, ε, εμεί ήμασταν τολμηροί, μπορέσαμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Στο θέμα των εξωτερικών υποθέσεων, να υπογραμμίσω ότι η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω παγκόσμιο παίκτη εξαρτάται από την ικανότητά μα να έχουμε μια επιτυχημένη πολιτική και από την ικανότητά μα να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας. Περιμένουμε από την Επιτροπή να είναι ε, ξεκάθαρη ως προς την προστασία του κράτους δικαίου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Και αυτό σημαίνει να αντισταθούμε στον Πούτιν, τον Ερντογάν, στον Μπολσονάρο, αλλά και στον Βίκτορ Όρμπαν, σε όλους αυτούς τους τύπους αυτού του κόσμου. Ε, θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουν οι συζητήσεις ένταξης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ε, κύριοι υποψήφοι επίτροποι, είναι πολύ σημαντικό να ε, εφαρμόσετε ένα σωστό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή με δίκαιη μετάβαση, να επιδιώξετε τους στόχους της χιλιετίας, καλύτερη προστασία για τους ε, εργαζόμενους. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι υπό την καθοδήγηση του κυρίου Τίμερμανς με μια ισχυρή ομάδα σοσιαλδημοκρατών επιτρόπων, αυτή η επιτροπή θα είναι κοντά στους πολίτες και θα είναι είναι έτοιμη να ακούσει και να αντιμετωπίσει με ενδιαφέρον τις ελπίδες τους και τις ανησυχίες τους. Για ένα λεπτό, η κυρία Ινφέλτε. Κυρία Πρόεδρε, εδώ είμαι, αν δεν με βλέπετε. Ε, έχω ντυθεί και στα πράσινα. Εγώ θα σας στηρίξω αλλά θα είναι ψήφος μου ψήφος πραγματισμού και όχι πάθους. Υπάρχουν αρκετά θετικά. Έχουμε πολλούς καλούς, εξαιρετικούς επιτρόπους, ε, τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γυναικών που υπήρξε ποτέ, το Πράσινο Σύμφωνο και ε, στιάζεται στην ε, γεωπολιτική. Αλλά θα είμαι ειλικρινή, ειλικρινής. Δεν θέλετε να αποσύρετε τον ε, επίμαχο τίτλο του χαρτοφυλακίου για τη μετανάστευση. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι τελικά ε, κατ' ουσίαν προβαίνεται σε μια ε, κοσμητική αλλαγή, αλλαγή εξοραϊσμού. Μέχρι τώρα, κατ' ουσίαν, είσαστε υποψήφιο των εθνικών κυβερνήσεων. Οι 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που σα ψήφισαν φέτο ε, δεν ψήφισαν για μια Ευρώπη που δουλεύει σε απομονωμένα δωμάτια, αλλά για μια διαφανή δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να καταδείξετε κατά πόσο ανήκετε στην παλιά ή στη νέα Ευρώπη. Ε, θα έχετε την ψήφου μου, τώρα πρέπει όμως και να επιτύχετε και τον ε, ενθουσιασμό μου. Για ένα λεπτό, ο κύριος ε, Ουρτουσάν, Ουρτασούν παρά την προσπάθεια που κάνατε εσείς ε, και, το συλλογικό, και συλλογικά επίτροποι, δεν θα σας υπερψηφίσουμε, κυρίως γιατί αφήσατε ε, την ε, πολιτική στα χέρια του Βίκτορ Όρμπαν. Όμως και το θέμα της, της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας ανησυχούν πάρα πολύ ως φεμινιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας, σας διαβεβαιώ ότι θα προσέχουμε σε κάθε βήμα που θα κάνετε σε αυτά τα χαρτοφυλάκια. Ωστόσο, κυρία Βαντελάιεν, δεν ήρθαμε για να είμαστε απλοί θεατές. Ε, δεν θα μείνουμε στην άκρη. Έχουμε έρθει εδώ για να αλλάξουμε τα πράγματα και για να δώσουμε νέα όθηση στο ευρωπαϊκό project. Θα δουλέψουμε σε τομεί όπως η εξωτερική πολιτική, θα ανταποκριθούμε στην, με σοφαρό τρόπο στη προβλήματα του κλίματος και εδώ θα βρείτε μια ομάδα ε, ευρωβουλευτών που είναι έτοιμοι να ε, ανασκουμποθούν και να δουλέψουν. Υπάρχουν δυσκολίε για να υπάρξουν πρόοδοι στο κοινωνικό στο περιβαλλοντικό και στο φεμινιστικό ε, τομέα που χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Ένα λεπτό, Βιλίμσκι. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που μου δίνετε το λόγο. Πολλοί από εσάς ε, χειροκροτούν αυτή την Επιτροπή. Εγώ διαφωνώ έχω αντίθετη άποψη. Ε, λάθος αυτή η Επιτροπή για δύο λόγους. Πρώτον, βλέπουμε ότι αυτή η Επιτροπή αποτελείται από 26-27 επιτρόπους ε, και θα πρέπει να περιστεί τουλάχιστον κατά ένα τρίτο για να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη, πιο εργατική. Ε, αυτός ο μεγάλος αριθμός των επιτρόπων συνεπάγεται και ένα πρόβλημα ότι τελικά ε, επειδή είναι πάρα πολλοί ε, και θέλουν να δείξουν στις πατρίδες τους ότι κάτι κάνουν και δεν είναι γνωστοί θα έχουμε πάρα πολλούς κανόνες, πολλές ρυθμίσεις όλα αυτά για να αιτιολογούν το αξίωμά τους. Ε, δεύτερον, δεν έχει επισημανθεί ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν μεγαλύτερο συγκεντρωτισμό και τους άλλους που θέλουν περισσότερη κυριαρχία των κρατών κρατών. Κανείς δεν τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό. Αλλά σας λέω το σημαντικότερο είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι ακριβώς χρειάζεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια στα σύνορα, μεγαλύτερη ευημερία και όχι στην ε, Ήπειρο αυτή να υπάρχουν όλο και περισσότεροι κανονισμοί. Ο κύριος Τέρτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω τους 13 ε, Γάλλους ε, φαντάρους που ε, έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα κατά του Ισλαμικού φονταμεταλισμού. Στη συνέχεια, κυρία Βαντελάιεν, θα σας πω ότι εμείς θα καταψηφίσουμε την Επιτροπή σας, διότι πιστεύουμε πως ε, ε, ξεκινάμε μια, ένα, μια ιδεολογική περιπέτεια που πραγματικά δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και τις διάφο τα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Ε, ούτε και τους τομείς που αυτή τη στιγμή φοβούνται πάρα πολύ γιατί όπως σας είπα ξεκινάτε μια περιπέτεια που όλος μας ανησυχεί αυτό δηλαδή που αποκαλείται Green Deal, πράσινο σύμφωνο είναι ένα όνειρο τρελό που βασίζεται σε απατηλές χήμερες και που απαιτεί όχι μόνο τεράστια ποσά που θα κινητοποιηθούν εδώ για να ελεγχθεί ακόμη περισσότερο το κράτος, να ελεγχθούν ακόμη περισσότερο τα κράτη ε, και οι επιχειρήσεις, ε, αντίθετα δηλαδή με τις ελευθερίες, ε, αλλά θα απαιτήσει και τεράστιες θυσίες από τα διάφορα κράτη και τους τομείς που δεν θα έχουν καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ευχαριστώ κύριος Παπαδάκη, σε ένα λεπτό η νέα επιτροπή διακρίνεται από τα ίδια αντιδραστικά υλικά που είναι φτιαγμένη και η ευρωπαϊκή ένωση αφοσίωση στην αντιλαϊκή πολιτική για ευέλικτη εργατική δύναμη ακόμα πιο φθηνή στα ελάχιστα κατεδάφιση κοινωνική ασφάλισης ψίχουλα στην ακραία φτώχεια χτύπημα τη συνδικαλιστική δράση, μαζικό φακέλωμα γενικευμένε απελάσει προσφύγων και μεταναστών. σε περίοδο ανεμική ανάκαμψη και με σημάδια στον ορίζοντα μια νέα, πιθανή συγχρονισμένη κρίση, προωθούνται τα πράσινα ταμεία και οι αδρές επιδοτήσεις για τα ψηφιακά μεγάλα πεδία κερδοφορίας των ομίλων και αυτά εν μέσω εμπορικών πολέμων αντιθέσεων και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ένωσης για τη στάση απέναντι σε ηπα κίνα και ρωσία την έκβαση του brexit την ένταση της στρατιωτικοποίησης. συμβολικό και ουσιαστικό ότι επικεφαλής της επιτροπής επιλέχθηκε η πρώην υπουργός πολέμου της γερμανίας. ανοίξατε και κλείσατε την ομιλία σας κυρία φοντερ με αντικομουνισμό δείχνοντας τον αντίπαλό σας φανερώνοντας αδυναμία και φόβο για την ιστορική αλήθεια και την πάλη των λαών που θα δυναμώσει ενάντια σε ευρωπαϊκή ένωση κεφάλαιο και κυβερνήσεις για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Κυρία Βαντερλάιν, θα δώσουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή σα γιατί συμμεριζόμαστε τα ίδια θέματα για τη μετανάστευση, για την ευελιξία, για το ρόλο τη βιομηχανία, την εσωτερική ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, τον αγώνα κατά του καρκίνου, την έρευνα, τη σχέση με τι ΗΠΑ. Άρα δηλαδή έχουμε το ίδιο πολιτικό όραμα, όχι το γραφειοκρατικό. Βέβαια θέλουμε όλα αυτά να ε, μεταφραστούν σε συγκεκριμένε επιλογέ και στον επόμενο προπολογισμό. Βεβαίω και θέλουμε την ε, τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην τιμωρήσουμε τη βιομηχανία και τη γεωργία. Η βιομηχανία είναι σημαντική και η έρευνα για να υπάρχουν νέε θέσει απασχόληση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει σωστή πολιτική ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι επιχειρήσει μα να ανταγωνίζονται όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Να προστατεύσουμε λοιπόν από τον αθέμητο ανταγωνισμό, να έχουμε μια σωστή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε του Κινέζου, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα προβλήματα με το dumping και κοινωνικά και κλιματικά, όχι μόνο εμπορικά. Δημιουργούν προβλήματα στο παραγωγικό μα σύστημα. Να είμαστε ε, προσεκτικοί και όσον αφορά τη γεωργία. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε περικοπέ γιατί η γεωργία παραμένει θεμελιώδη στοιχείο για την προστασία του περιβάλλοντο, την αντιμετώπιση τη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και όσον αφορά τη μετανάστευση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προσέξουμε την Αφρική. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο μεγάλο πρόγραμμα Marshall για να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροέ προ την Ευρώπη. Και κάτι άλλο που αφορά το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό, αυτό που έκανε η Ντάφνε Γκαλίτσια, η δημοσιογράφος, να ε, συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό και ευτυχώς είμαστε πολύ κοντά στο να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Για 1,5 λεπτό η κυρία Φρίτσον. Σήμερα είναι σημαντική μέρα, κυρία Πρόεδρε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εγκρίνουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία και νομίζω ότι είναι σημαντικός στόχος η Ευρώπη να είναι η πρώτη ε, ήπειρο που θα είναι ουδέτερη από πλευρά άνθρακα. Το πράσινο σύμφωνο είναι πολύ σημαντικό, ώστε όλοι μαζί να υπομισθούμε τις ευθύνε μας και να αφήσουμε στα παιδιά μας μια βιώσιμη Ευρώπη και ένα πιο βιώσιμο κόσμο για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη μετάβαση. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερες δουλειές στην Ευρώπη και δουλειές με καλές συνθήκες απασχόλησης. Κυρίως για τους νέους της Ευρώπης. Ένα τρίτο των νέων είναι στην ανεργία. Τα κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να ενισχυθούν στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες επί του κοινωνικού πυλώνα, κάτι που υποστηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα πρέπει γρήγορα να βρούμε και μια μεταναστευτική πολιτική που θα είναι υπεύθυνη και αλληλέγγυα, όλοι μαζί. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε τη Γίλα Ιόανσον που είναι η γυναίκα που μπορεί αυτό να το πετύχει. Επίσης, καλωσορίζω την πρωτοβουλία της Επιτρόπου να έχουμε μια ισότητα στην Ένωση και μια ε, συγκεκριμένη ε, πολιτική για την ισότητα. Θέλουμε να προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, τα δημοκρατικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων και να δώσουμε αποτελέσματα στην προσπάθεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάουτμαντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε, κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, πεπισμένη θα ψηφίσω ναι. Ποτέ δεν είχαμε επιτροπή που να έχει τόσο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, που να έχει τόσες πολλές γυναίκες, ε, που να είναι τόσο φιλόδοξη σε θέματα σύλλου, μετανάστευσης ε, και άμυνας. Ενδιαφέρεται για την καινοτομία, την ψηφιοποίηση της οικονομίας μας. Ο κύριος Μπορέλ θα αγωνιστεί για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και εγώ θέλω να πιστεύω ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια διάσκεψη χωρίς σύνορα. Θα εξεταστούν πάρα πολλά θέματα, μεταξύ άλλων το ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης. Κυρία Φοντερ Λάιεν, ε, το μήνυμα είναι σημαντικό για μας. Ε, το ότι θα υπάρξει μια διάσκεψη για το πώς θα λειτουργεί η Ευρώπη στο μέλλον ε, προς όφελος του πολίτη. Και κύριε Βαντελάν, δεν θα σε εκπλήξει που θα σας προσφωνήσω ως Αμαζόνα. Μια Αμαζόνα που θα πάρει τα ενία στα χέρια της και θα οδηγήσει το άλογο της Ευρώπης στο σωστό δρόμο. Θα τραβήξετε την ενία, θα τρέξετε γκαλόπ με γρήγορο ρυθμό. Αυτά περιμένω από εσάς, ε, κυρία ε, Φοντελάν. Αν δεν τα κάνετε βέβαια αυτά, εμείς θα πάρουμε το μαστίγιο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς θα έχετε τραβήξει καλά τα ενία και θα συνεχίσετε να τρέχετε με γρήγορο ρυθμό. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, βλέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω αμφιβολίες κατά πόσο θα δράσει σύμφωνα με τα συμφέροντα των πολιτών, κατά πόσο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να χάσουν ε, την ταυτότητά τους και να υπακούν σε εντολές που έρχονται από μακρινό κέντρο. Βλέποντας για το, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν μας νοιάζει αν καίγονται τα δάση της Βραζιλίας ή κατά πόσο μέσω του Μερκοσούρ μεταφέρεται, εισάγεται βόλιο κρέας εδώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το χαρτοφυλάκιο της ε, κυρίας Γιούροβα προβληματίζει. Ε, Δίκαι, δικαιοσύνη, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ελευθερία, μη διάκριση, ανοχή, όλα αυτά Πώς αυτά μπορεί να ευθυγραμμιστούν με τεράστιες διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τις επιδοτήσεις που δίνονται για τη γεωργία και χώρες που δεν στέλνουν ευρωβουλευτές. Αυτές οι δικαιολογίε που προβάλλονται δείχνουν ότι τελικά γίνεται πραγματικότητα αυτό που περιέγραφε ο George Orwell τελικά στα δίγημά του. Αγαπητή κυρία Βοντελάιν, υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία διαφωνώ για την υφέρπουσα ομοσπονδιοποίηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται υπερκράτος και απογοητεύομαι ότι μετά από 40 χρόνια που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταφέραμε να σας πείσουμε ότι η επιτυχία της Ευρώπης εξαρτάται από την προστασία της κυριαρχίας των κρατών μελών. Αλλά σίγουρα θα αποχωρήσουμε. Και θέλω να σας πω ότι παρά τις διαφορές μας η Ευρώπη δεν έχει μεγαλύτερο φίλο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αναγνωρίζουμε τι προτεραιότητε για την αλλαγή του κλίματο, για την οικονομική ανταγωνιστικότητα, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και το κράτος δικαίου. Και δεν θα βρείτε μεγαλύτερο σύμμαχο από το Ηνωμένο Βασίλειο προ την επίτευξη των αμοιβαίων μα στόχων στους τομεί αυτού. Στο μέλλον θα έχουμε μεγάλα προβλήματα για να καθορίσουμε εκ νέου τη σχέση μα. Ελπίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θυμάται ότι ένα ελεύθερο, ισχυρό Ηνωμένο Βασίλειο που εμπορεύεται ελεύθερα ήταν πάντα προ το καλύτερο συμφέρον των Ευρωπαίων όπω και για τους ε, υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να πω ότι για το σύντομο διάστημα που είναι ευρωβουλευτή, ε, απόλαυσα και τη συντροφιά και τα επιχειρήματα των ε, συναδέλφων μου των ευρωβουλευτών. Προσβλέπω να συνεργαστώ μαζί σα και στο μέλλον που θα επιδιώξουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλου του ε, πολίτε μα. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Ρανζέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ομιλία που κάνατε, για το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε και για την ομάδα που συστήσατε και να σας ευχαριστήσω για την έμπνευση που μας δώσατε. Δώσατε σε ένα σωρό Ευρωπαίους και κυρίως εμάς που είμαστε εδώ σε αυτό το σώμα. Και γι' αυτό μπορώ να πω, αντίθετα από την Ολλανδέζα συνάδελφο, ότι μπορείτε να βασίζεστε στο ψήφο μου και στον ενθουσιασμό μου. Θα ήθελα να σας πω το εξή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον, τον προϋπολογισμό που να είναι μικρότερος από τον προηγούμενο και κυρίως πρέπει να δούμε τις πολιτικές συνοχής γιατί σήμερα υπάρχει μια απειλή ενάντια στη συνοχή και χωρίς συνοχή δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστήνω λοιπόν την προσοχή στο κίνδυνο του να σταματήσει να γίνεται κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, όπου έχουμε 5 εκατομμύρια για αυτά τα ζητήματα. Νέες προτεραιότητες σημαίνει νέα χρηματοδότηση. Η πολιτική συνοχή όμως δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Τέλος, να μου αφήσετε να πω κάτι για τη διάσκεψη για το μέλλον για την Ευρώπη. Πιστεύω πως δεσμευόμαστε σοβαρά ε, εάν θα πρέπει να είμαστε ικανοί να εμπλέξουμε τους πολίτες και αν η Κομισιόν δεν κάνει αυτή την προσπάθεια να μην φτιάξει περάσματα πριν ακριβώ να ακούσει του ίδιου του πολίτε. Πιστεύω πω αυτά είναι βήματα σημαντικά για αυτή την Επιτροπή και για του θεσμού να κάνουμε μια διάσκεψη επιτυχή για το μέλλον τη Ευρώπη. 1,5 λεπτό ο κύριος Μωράης τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι Βρετανικές εκλογές δεν ε, αποκλείουν το να στείλουμε Βρετανό Επίτροπο. Είναι νομική μας υποχρέωση και είναι ένα λυπηρό ζήτημα γιατί η, η ειλικρινή συνεργασία είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ ε, και δεν είστε νομικός πλήρης και αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτός είναι και ο λόγος Βλέπουμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα ε, δεν έχει ασχοληθεί με θέματα όπως η μείωση των εκπομπών, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όλα αυτά έχουν πλέον χαρακτηριστεί από καθυστερήσεις και από προκλήσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξει μια πιο προοδευτική επιτροπή και γι' αυτό ψηφίσαμε προς την κατεύθυνση αυτή να πω κάτι το οποίο το λέω συνέχεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ένα ήταν οι 39 μετανάστες μέσα στο φορτηγό και από την άλλη οι άνθρωποι που πνίγονται στη Μεσόγειο. Λοιπόν, υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις αυτή τη στιγμή ξεκινήσετε τη δουλειά σας. Η πρόκληση είναι πράγματι τεράστια, είναι θηριώδης Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και η δραστηριότητά σας ήθε να σέβεται πάντα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τα θεμελιώδη δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Εμείς δεν θέλουμε ε, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες να είναι στην απέναντι πλευρά εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί δίκαια στη διεθνή σκηνή. Ο κύριος Μπέρνς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι οι επίτροποι έχουν υψηλή ποιότητα. Αναφέρομαι και στον Νικόλα Σμίτο, του οποίου η αρμοδιότητα δεν αμφισβητείται από κανέναν. Απ' την άλλη δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τη, τη Σιλβί η οποία ήταν εξαιρετική υποψήφια, αλλά η οποία δεν αντιμετωπίστηκε σωστά κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της ακροάσεως. Προφανώς η ακρόαση δεν είναι κάτι το ευχάριστο και ε, μπορεί να τεθούν και είναι επιθυμητό. Δύσκολες ερωτήσεις, είναι απαραίτητο. Πέραν τούτου όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται ή ε, γεμάτη έλλειψη αντικειμενικότητας, επιθετικότητα και μίσος. Και είχαν πει πριν την ε, ακρόαση κάποιοι «We will kill her». Σε τέτοιο στάδιο έφτασαν. Γι' αυτό λοιπόν όταν λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο στην ουσία τι κάναμε, διώξαμε ένα εξαιρετικό ταλέντο. Δεν μπορώ να αποδεχθώ την απόφαση αυτή και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη. Μαντίσον, ένα λεπτό. Δυστυχώς είναι αδύνατο να υποστηρίξουμε αυτή την Επιτροπή γιατί διότι της λείπει ε, δημοκρατική νομιμότητα. Η κυρία Βαντερ Λάιεν δεν ψηφίστηκε από τις ευρωεκλογές Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε φυσικά, αλλά θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αν είχε εκλεγεί, αλλά δεν εξελέγει. Θα είχαμε ε, καταλάβει, θα είχαμε ε, ε, συμφωνήσει αν είχε καλύτερε ικανότητε, ωστόσο όχι. Για παράδειγμα, παρακολουθείτε από το γερμανικό κράτος για διάφορους λόγους. Με αυτή τη νέα Επίτροπο στην κορυφή το μέλλον της Ευρώπης φαίνεται σκοτεινό. Δυστυχώς αυτή η Επιτροπή δεν νομίζουμε ότι θα μπορέσει να μας δώσει ένα φωτεινό μέλλον. Η ιστερία τώρα για το κλίμα και η μάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, για το εμπόριο μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Είναι ελεύθερη η συμμετοχή των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μάντισον, υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρα. Τη δέχεστε. Ζητώ συγγνώμη, κύριε. Ο κύριο Κάρα, όχι, δεν ζήτησε ε, μπλε κάρτα, ζήτησε catch Εντάξει, λοιπόν. Να πω ότι η διαδικασία catch έκλεισε πριν λίγο, διότι έχουμε μεγάλο κατάλογο. Επόμενο ομιλητή για μισό λεπτό, η κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ. Αντίθετα με τον προλαλήσαντα, εγώ πιστεύω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξίζει τη στήριξή μας και την εμπιστοσύνη μας. Και αναφέρθηκε στη Βελούδινη Επανάσταση και τον Βάκλαπ Χάβελ η κυρία Φοντερ Λάιεν. Εφόσον εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, ε, σημαίνει ότι μπορεί να αναλάβει το έργο της και να δουλέψει για τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας οι συντονιστές, ε, μιλάω εκ μέρους των συντονιστών της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και πρέπει να τονίσω ότι η εκλεγμένη πρόεδρος ε, συμπλήρωσε το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Γκάμπριελ με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και ακόμα και για την υγεία δεν είναι βέβαια ο αθλητισμός στο χαρτοφυλάκιο αυτός καθεαυτός, γι' αυτό να εγκρίνεται μια δικαινοβουλευτική ομάδα που να ασχολείται με τον αθλητισμό έτσι ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί ιδιαίτερα και με τον αθλητισμό. Και ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση να στηρίξει το τριπλασιασμό του προπολογισμού για το πρόγραμμα Έρασμο, το οποίο έχει τεράστια προστιθέμενη αξία. Ε, βοηθάει δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους. Είναι μια τεράστια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Βοηθάει την ε, συμμετοχή όλων και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Επίσης, να ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης για τους εθελοντές, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τους Ευρωπαίους. Ευχαριστούμε ο κύριος Κούμπουλος. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας συγχαρώ για όσα είπατε μέχρι τώρα κύριε Φοντερ και για αυτά τα οποία θα κάνετε. Είσαστε γυναίκα με πολιτική εμπειρία. Σας εμπιστεύομαι. Δεν ε, σκοπεύω να σας δώσω περισσότερες πολιτικές συμβουλές, έχετε ήδη πάρει αρκετές. Είπατε τι σκοπεύετε να πετύχετε και είναι ένα τεράστιο άθλος εφόσον τα καταφέρετε. Θέλω να σας ευχηθώ να μην χάσετε τον προσωπικό σας ενθουσιασμό, την ενέργειά σας, τις ηγετικές σας ικανότητες. Ε, κάτω από δύσκολε συνθήκε. Έχω πέρασει και εγώ από κρίση και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα τότε. Πριν από μερικά χρόνια. Να ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει εσάς προσωπικά και την Επιτροπή σας, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές μας χωρίζουν. Να κάνουμε τη δουλειά μας, να ζήσουμε απλά και να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλή τύχη. Ευχαριστούμε. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή να τηρείτε το ένα λεπτό για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι αγορητές. Η κυρία Σπυράκη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Φοντερ Λάιεν, Πρόεδρε της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ψήφος μας που σας δίνουμε σήμερα είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Πράσινη Συμφωνία που μπορεί να αποτελέσει την αιτία για την αλλαγή της οικονομίας και της ζωής μας στην ευρωπαϊκή ένωση αρκεί να συμφωνήσουμε εδώ ότι χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ενθάρρυνση με όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε για την καινοτομία μαζί με την ευρώπη που θα πάει μπροστά που θα είναι η πρώτη ήπειρος με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το 2050 υπάρχει όμως και η ευρώπη που εξαρτάται από τον άνθρακα και δεν πρέπει να μείνει πίσω οι χιλιάδες οικογένειες στις 41 μία που εξαρτώνται από τον άνθρακα στη δυτική μακεδονία στη μεγαλόπολη περιμένουν από εσάς σήμερα να υποστηριχθούν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι θα έχουν πολλές και βιώσιμες δουλειές στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν. η δίκαιη μετάβαση που θα βασιστεί στο ταμείο δίκαιης μετάβασης οφείλει να είναι στην κορυφή της ατζέντας σας. σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Μπέρλι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα υποστηρίξω ολόκληρη την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι δεν συμφωνώ απόλυτα. τους ε, περασμένους μήνες ε, είχαμε μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Σλοβενία και εύχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλή τύχη. Έχετε μεγάλες προκλήσεις μπροστά σας. Οι μετασχηματισμοί στο κοινωνικό τομέα, στο πράσινο τομέα, στον ψηφιακό τομέα, μαζί με μια δίκαιη μετάβαση, είναι μεγάλες προκλήσεις. Θα πρέπει να μην αφήσουμε κανένα πίσω, να έχουμε υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι συνολικές τεχνικές εξελίξεις και οι επενδύσεις ε, ε, και ε, στις υποδομές, η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν, όπως επίσης και η πολυμορφία και το διεθνές δίκαιο. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ο κύριος Χόουαρντ. Είπατε ότι είσαστε Remainer, υπέρ ε, δηλαδή τη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ λοιπόν, και πολύ χαίρομαι για τα λόγια σα αυτά. Τώρα λοιπόν ολοκληρώνουμε μια διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να ψηφίσουμε υπέρ τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αρχίσει να εργάζεται ε, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει μα, η κλιματική αλλαγή, αδικίε, ε, διακρίσει κλπ. Να ξέρετε ότι και εγώ θλίβομαι που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παραβεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν έχει ορίσει επίτροπο. Οι υπόλοιπε 27 χώρες έχουν διάφορα χαρτοφυλάκια ε, τα οποία έχουν αναθέσει στους καλύτερους της Ευρώπης. Η δικιά μας κυβέρνηση αποφάσισε να αφήσει τη δικιά μας θέση κενή. Να λοιπόν ένα παράδειγμα στην ιστορία ενός έθνους που δουλεύει για να έχει λιγότερη επιρροή, για να έχει λιγό... χαμηλότερη φωνή και στο τέλος να σιωπά. Δεν έχει και πολύ νόημα. Θα ήθελα περισσότερη λογική. Ευχαριστούμε, κυρία Τόμασιτς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ η καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το οργανωτικό πλαίσιο, κάποιοι νέοι τίτλοι επιτρόπων και κάποια νέα χαρτοφυλάκια δημιουργούν κάποια επίπεδα σύγχυσης. Η προηγούμενη αυστηρά τεχνοκρατική, αν θέλετε, μορφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αντικατασταθεί από μια ιδεολογικοποιημένη, αν θέλετε, ε, άρθρωση πλέον. Οι συμφωνίες έγιναν ανάμεσα στα κράτη-μέλη και εξυπηρετούν τις πολιτικές τους σκοπιμότητες. Σας ψηφίσαμε κυρία Φόντερ Λάιεν για λόγους πραγματισμού, ελπίζω να ανταποκριθείτε. Φερέιρα. Πρόεδρε. Ε, για το πολιτικό σας πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι έχετε σαν ε, βασικό στόχο την πρόθεση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ουσία θέλετε να επενδύσετε ακόμα περισσότερο στην απόλυτη κυριαρχία ε, της ενιαίας αγοράς εις βάρος των χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικά θέματα εξυπηρετείτε το μεγάλο κεφάλαιο, εξυπηρετείτε τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κυριαρχούν στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η πολιτική συνοχή υπόκειται πλέον σε αυτό που ονομάζουμε διαρθρωτική πολιτική που σημαίνει την προσωρινή απασχόληση και κυρίως την διάλυση του δημόσιου τομέα και αυτό φαίνεται και από την κατανομή των χαρτοφυλακίων σας. Υπάρχει μια σαφή στροφή προς τα δεξιά και η αντίθεση ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες οξύνεται όλο και περισσότερο. Πρόεδρε Ούρσουλα, εγώ πολιτικά σας υποστηρίζω, όπως και όλη την Επιτροπή και σα καλωσορίζουμε για την επόμενη πενταετία, ειδικότερα οι συνάδελφοί μου από την, τον συνάδελφό μου από την Ιρλανδία, τον κύριο Χόγκαν. Σας, ε, βλέπουμε πως ε, χτίσατε υποστήριξη για την υποψηφιότητά σας και πως καταφέρατε ε, και την υποστήριξη είχατε καταφέρει την υποστήριξη των πρασίνων που αποτελούν το 10% του Κοινοβουλίου. Ε, δεδομένου όμω ότι τελικά δεν θα σα υποστηρίξουν σήμερα και μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι με οτιδήποτε ε, κάνετε εσεί με τη Νέα Πράσινη Συμφωνία, όσο φιλοδοξή και αν είναι, εσεί και ο κύριο Τίμερμαντ μπορεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αλλάξετε τον τίτλο σε μια ενισχυμένη κλιματική στρατηγική για την Ευρώπη. Αυτό που θα είναι πραγματικά δηλαδή, διότι όλοι ε, όλα τα πολιτικά κόμματα δεσμευόμαστε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ανομάζοντα την ενισχυμένη κλιματική στρατηγική, θα μπορούσατε να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μάρκο. Ναι, ε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής. Ε, πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά. Έχετε την υποστήριξη της πολιτικής ομάδας μας, διότι υιοθετήσατε τις προτάσεις μας και έχετε κάποιους από τους καλύτερους ε, μεταξύ ημών στην ομάδα σας. Ωστόσο δεν πρέπει να παραμένουμε στα ωραία λόγια, πρέπει να υλοποιηθούν και να υπάρξουν επαρκή κονδύλια. Πρέπει να εστιαστούμε στο μέλλον της Ευρώπης. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν θα περιμένουν ενώ εμείς κολυσιεργούμε. Ε, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Πλημμύρες, ε, οι καταιγίδε, η Κίνα και η ΙΠΑ ε, δεν διστάζουν όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση. Ωστόσο, ένα σωρό φτωχοί άνθρωποι πεθαίνουν. Δεν, μπορούμε, δεν έχουμε περιθώριο για διαφορία. Έχει έρθει η ώρα να δράσετε και θα έχετε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου αυτού για τις πρωτοβουλίες σας. Να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το Εθνικιστικό Βασικό Κόμμα υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει εξίσου άντρε και γυναίκε και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία. Μα ενδιαφέρουν οι αξίε, όχι τα συμφέροντα. Μια βιομηχανική πολιτική ισχυρή υπέρ του παραγωγικού τομέα και η αλλαγή του παραγωγικού μας ε, μοντέλου. Επίσης, το ότι επήγει το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να στοιχηματίσουμε στη βιωσιμότητα, αλλά και να εξαρτήσουμε την οικονομία μας από την παραγωγή. Κοινωνική προστασία επίσης, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αξιοπρεπή έσοδα και μια ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις περιφέρειες και τους δήμους που υποδέχονται μετανάστες. Έπειτα, το μέσο για να ελέγχεται το κράτος δικαίου δεν θέλουμε αυτού που θέλουν ε, να μα πάνε πίσω. Περισσότερη δημοκρατία θέλουμε. Δημοκρατία με κεφαλαίο, συμφωνίες, ανθρωπισμό. Θέλουμε... Διακόπτη πρόεδρο. Ο κύριος Παπαδημούλης, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Φόρντερ Λάιεν, θα καταψηφίσω τη νέα Κομισιόν και το πρόγραμμά της, γιατί πιστεύω ότι οι στόχοι που θέσατε είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν με έναν προϋπολογισμό μόνο 1% του ευρωπαϊκού αεπ γιατί διαφωνώ με τις περικοπές τις μεγάλες που κάνει η κομισιόν στις πολιτικές για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική γιατί θεωρώ ντροπή η ευρωπαϊκή ένωση να έχει παραλύσει και να μην μπορεί να δώσει μια ευρωπαϊκή απάντηση στηριγμένη στην ανθρωπιά και στο κράτος δικαίου στο θέμα το προσφυγικό γιατί δεν θέλω η κομισιόν να είναι όμηρος των κυρίων όρμπαν και σαλβίνη και γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξους στόχους και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας. γι' αυτό η ευρωομάδα της αριστεράς θα καταψηφίσει τη νέα κομισιόν και θα ασκεί επικοδομητική αυστηρή αντιπολίτευση κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αξιότιμη Επιτροπή, θα ήθελα να σας ε, ε, συγχαρώ κυρία Βεντελάν, για την εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που υπάρχει σε εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και πιστεύω ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία και αποτελεσματική. Έχετε τις σωστές ε, προτεραιότητες. Υγεία, ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και οι στόχοι ε, και τα μέτρα πρέπει να υποστηρίζονται και από τον προϋπολογισμό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά τους στόχους αυτούς. Αυτό που με χαροποιεί περισσότερο είναι ότι στο επίκεντρο των πολιτικών σας έχετε θέσει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο με τις ανάγκες του. Εμείς ε, στην Ευρώπη παντού έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Ασφάλεια, ειρήνη, συνεργασία. Αυτές είναι οι αξίες που έκαναν την Ευρώπη μεγάλη. Ευχαριστούμε κύριο Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι αποφάσισε να παρουσιάσει σχέδιο δύο οδηγιών με στόχο να εισάγει φόρο στα έσοδα από διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες. Επίσης, εσείς, κυρία Φοντερ Λάιεν, αναφέρατε ένα πράγμα, δίκαιο ψηφιακό φόρο. Εγώ θέλω να εκφράσω την απόλυτη στήριξή μου για ένα τέτοιο μέτρο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία υλοποιώντας τους στόχους αυτούς που πιστεύω ότι είναι πολύ βασικοί. Δυστυχώς ξέρω ότι οι εργασίες στο Συμβούλιο δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η εισαγωγή ενός τέτοιου ψηφιακού φόρου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αντιστέκονται, που είναι κατά. Παρόλα όλα αυτά όμως, ε, κυρία Πρόεδρε, σας εύχομαι να αντισταθείτε εσείς από τη δικιά σας την πλευρά και να συνεχίσετε να δουλεύετε με συνοχή και να μην αποσύρετε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Φοντερ Λάιαν, έχετε την υποστήριξή μας και σας συγχαίρω για την πολύ ε, ικανή και εξισορροπημένη ομάδα έχετε αναφέρει τα σωστά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την ψηφιοποίηση, την υγεία, τα δημογραφικά προβλήματα. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι θέλετε να επιλύσετε τα προβλήματα έτσι ώστε να δημιουργήσετε νέε ευκαιρίε. Και αυτό θα αποτελέσει την εγγύηση ότι η Ευρώπη θα γίνει ομορφότερη ε, ήπειρος ε, του κόσμου ε, θα παραμείνει η ωραιότερη ήπειρος του κόσμου όπου ο κόσμος ζει με μεγάλη ευχαρίστηση και την αγαπά. Χαίρομαι που η διεύρυνση ε, τη Ευρώπη προ τα Δυτικά Βαλκάνια έχει τη δική σα υποστήριξη. Πρέπει να βοηθήσουμε να εκδημοκρατιστούν όλα αυτά τα κράτη και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε να καλύψουν το χαμένο έδαφο σε θέματα ανάπτυξη αλλά και τα δημογραφικά προβλήματα. Είναι ένα πρόβλημα. Η ε, ε, κυρία Γκραπίνη. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Εκλεγμένη Πρόεδρε, θέλω να πω ευθύ εξ αρχή ότι εγώ σα ψήφισα και παρακολούθησα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε σήμερα. Ε, πρέπει να απαντήσετε σε πολλέ ερωτήσει. Εγώ θα ήθελα να ε, τονίσω το θέμα της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Παραμένουν τρεις χώρες μέλη που δεν συμμετέχουν στο χώρο Σέγγεν. Εγώ θα ήθελα εσείς να απαντήσετε και γι' αυτό, δηλαδή για τις αρνητικές πτυχές. Δεν θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα και να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Τα κλεμμένα παιδιά, η βία σε βάρος των γυναικών, η ανάμεξη στις εκλογές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν οδηγήσει στη μείωση της εμπιστοσύνης του κόσμου. Εμείς πρέπει να ξέρετε ότι θεωρούμε τη σημερινή ψηφοφορία πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να βοηθήσει να ε, έχουμε και πάλι εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκλεγμένη πρόεδρο, κύριε Λάιεν και διακόπτουμε μέχρι τις 12 ακριβώς. Presidente. Ah, riecco, rieccoci. Eh? Prendiamo posto, colleghe, colleghi. Καθίστε παρακαλώ. Innanzitutto vorrei dare θα ήθελα να καλωσορίσω Συνάδελφοι, ακούστε με λίγο. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε συνάδελφοι. Θέλω να καλωσορίσουμε στα τιμητικά θεωρία ε, τους εκπροσώπους ε, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής των Συμβούλων της Ιαπωνίας. Τους καλωσορίζουμε. Βρίσκονται εδώ για την διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας πρόεδρος της αντιπροσωπείας, εκπρόσωπος της δίαιτας της Ιαπωνικής είναι ο, ο κύριος Όνο Ντέρα. Τους καλωσορίζουμε στο Στρασβούργο. Να καλωσορίσω επίσης πάντα στα ίδια θεωρία 80 μαθητές που συνοδεύονται από τους καθηγητές τους που ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρουσιάσουν την δήλωσή τους για τα δικαιώματα του πλανήτη. Τους καλωσορίζουμε. Σας καλωσορίζουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. E e λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με τις ψηφοφορίες για την εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και δύο μέρες 13 Γάλλοι στρατιωτικοί έχασαν την ζωή τους στα πλαίσια μιας επιχείρησης εναντίον της τρομοκρατίας και το Κοινοβούλιο δεν τήρησε ενός λεπτού σιγή για να τους τιμήσει. Γι' αυτό σας προτείνω ακριβώς αυτό και όλοι οι συνάδελφοι να σηκωθούν για τους στρατιώτες της Ευρώπης που θυσιάστηκαν στο Μαλί. Για μια στιγμή παρακαλώ. Κύριε Ζαντό, Ίσως εσείς δεν ήσασταν παρόν χθε στην Ολομέλεια, διότι ακριβώς αποτίσαμε φόρο τιμής στους στρατιωτικούς αυτούς. Ίσως να ήσασταν αφηρημένους, ίσως να ήσασταν απόν. Αλλά εμείς ήδη τιμήσαμε τους στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στο Μαλί. Αλλά δεν θα σας δώσω το λόγο πάλι, αλλά θα ήθελα να πω μιας ε, και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι κοινό αίσθημα όλων των κοινοβουλευτικών, εγώ σας προσκαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Iniziamo. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία για την εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας ενημερώσω ότι θα προηγηθεί μια παρέμβαση από πλευρά των πολιτικών ομάδων αντίστροφα. Ο κύριος Φόξ έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας είμαστε ειλικρινεί με τους ψηφοφόρους μας. Η διαδικασία αυτή είναι γελία. Εμείς είμαστε σαν ε, ε, μια σκιώδης ε, στρατιωτική δύναμη που έρχεται δίθεν να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Το κοινοβούλιο αυτό είναι μια σκέτη δημοκρατική κοροϊδία ε, και δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ε, μορφές λήψης απόφασης. Κάναμε κάτι αστείες, ε, ψευδεπίγραφες ακροάσεις και δεν έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε πραγματικά. Πρόκειται για κάτι το υποκριτικό. και αυτό χαρακτηρίζεται και από το τεράστιο πόστερ ε, της Φόντερ Λάιεν έξω από το κτίριο στο στρασ στις Βρυξέλλες ήδη. Στις Βρετανικές εκλογές ε, που θα γίνουν τότε θα ζήσουμε μια πραγματική στιγμή δημοκρατίας. Η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσει ε, δεν αρκούν δεν ψήφισε ο λαός την κυρία Φόντερ Λάιεν. Ε, στους διαδρόμους έγιναν συζητήσεις παρασκηνιακές και κατέληξαν σε μια μορφή συμβιβασμού και τώρα θα έχει τη δύναμη να προτείνει την πολιτική της Ευρώπης που θα επηρεάσει τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών είτε τους αρέσει είτε όχι. Το Green Deal, η λιτότητα, και μάλιστα με ανθρώπους μαζί της όπως ο Γιώση Μπορέλ που ξέρουμε πώς ακριβώς ε, σκοπεύει να ασκήσει πολιτική. Όλα αυτά στην ουσία είναι μια κλοπή της δημοκρατίας από τα χέρια του λαού. Εμείς λοιπόν δεν θα συνενέσουμε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ψηφίζουμε σε λίγες μέρες και θα επιλέξουν την κυβέρνησή τους οι Βρετανοί. Σας ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, συνεχίζει η κυρία Φόξ. Ε, οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ποια είναι η πραγματική δημοκρατία. Κυρία Ομπρί, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Η σημερινή ψηφοφορία δεν μοιάζει με τις άλλες. Είναι πάρα πολύ σημαντική ίσως η ψηφοφορία του αιώνα για να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, την κλιματική καταστροφή και την κρίση των ανισοτήτων. Δύο διακυβεύματα που δεν ε, μπορούν ε, να βασιστούν σε δεσμεύσεις ε, αντιφατικές. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να διαπιστώσουμε ότι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στους στόχους μας. Τρεις ε, τροπή απομακρύνθηκαν λόγω συγκρούσει συμφερόντων. Ε, και υπάρχουν και αφιβολίε και για άλλα μέλη τη Κομισιόν. Φυσικά, επί τη ουσία υπάρχουν διάφορε υποσχέσει. Ε, πολύ καλέ τα ελάχιστο εισόδημα και διάφορα άλλα. Για όλα τα θέματα αυτά θα μας έχετε ως συμμάχους που θα σας παρακολουθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Ωστόσο, πέραν αυτών παραμένετε σε δόγματα που δημιουργούν κοινωνική κρίση και άλλα προβλήματα σήμερα. Πώς θα προωθήσετε το Green Deal, πώς θα καταπολεμήσετε τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή ενώ υποστηρίζετε τους χειρότερους φορολογικούς παραδείσους, πώς υποστηρίζετε μια ανθρωπιστική πολιτική και πώς θα δώσετε ελπίδα στους ευρωπαϊκούς λαούς ε, ενώ συνεχίζετε η λιτότητα. Δεν μπορείτε να είστε αυτοί που υποστηρίζετε τους λαούς ε, και ταυτόχρονα να κάνετε άλλα. Σήμερα ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, την επιφυλακτικότητα των πολιτών προς τα ευρωπαϊκά όργανα που ο πλανήτης χρειάζεται ένα νέο φιλόδοξο Green Deal να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις υποστηρίζοντας τη γεωργία, της βιομηχανικές μας πρακτικές, ε, το, τρόπους κατανάλωσής μας χρειαζόμαστε φορολογική δικαιοσύνη να πάψουν να μένουν ατιμόρυτες οι πολυεθνικές που δεν καταβάλουν